σύμφωνα με το άρθρο 135 του κανονισμού θα κρατήσει η συζήτηση αυτή μια ώρα. Το πρώτο λοιπόν από αυτά τα θέματα είναι το σχέδιο ψηφίσματος για το Μπουρούντι και την υπόθεση του Μπομπ Ρουγκουρίκα. Δίνω τον λόγο στην κυρία Σαρτζεντίνη για, ε, να, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο Μπομπ Ρουγκουρίκα είναι δημοσιογράφος από το Μπουρούντι, διευθυντής του Ράδιο Αφρίκα. Στις 20 Σεπτεμβρίου φυλακίστηκε για... γιατί έδωσε κάποιες ε, πληροφορίες για την δολοφονία τριών Ιταλιδών, ε, Ιταλίδων καλοβρέων. και τώρα ε, είναι στη φυλακή γιατί πολύ απλά ε, έφερε σε δύσκολη θέση την εξουσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ζητάει την άμεση απελευθέρωση του Μπομπ Ρουγκουρίκα γιατί πρόκειται για μια προσπάθεια φήμωσής του. Αυτό πρέπει να το δούμε βεβαίω και υπό το φως των επερχόμενων εκλογών στο Μπουρούντι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό Ρίτσαρντ Τσαρνέτσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε. Θα πρέπει να δούμε ότι πρόκειται για αλληλεγγύη, πρόκειται για τη στοιχειώδη δικαιοσύνη που πρέπει να επιδείξουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τα πρόσωπα αυτά που βρίσκονται σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Η εξουσία διώκει κάποιον ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του σαν δημοσιογράφος. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Τρεις Καλό είχε να σκοτωθεί και έκανε το καθήκον του αυτός ο δημοσιογράφος. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την πηγή του. Μα είναι κάτι σαν τον ιερέα σε σχέση με την εξομολόγηση. Δεν είναι δυνατόν να αποκαλύπτεται το περιεχόμενο της εξομολογήσεως. Πρόκειται επομένω για έναν καλό σκοπό και είναι σωστό το Πανεσκλητό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Επίσης ο επόμενος ε, συντάκτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε 432 εκατομμύρια. Τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Μπουρούντι για να βελτιώσει την διακυβέρνηση και τα της κοινωνίας των πολιτών. Όμως, από 160 θέσεις βρίσκεται στη θέση 142 η χώρα αυτή όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Σύμφωνα με, την, ε, με τον φορέα δημοσιογράφη χωρίς σύνορα. Μα δεν υπάρχουν ελεύθερες εκλογές αν δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος. Και επομένως είναι αφόρητο αυτό το οποίο γίνεται εδώ με τον κύριο Ρουγκουρίκα. 432 εκατομμύρια δώσαμε ε, και αυτό είναι αντιφατικό. Οπότε πέρα από τις ανησυχίες τις μεταφυσικές, τις ε, φιλοσοφικές, ε, όλα όλα αυτά τα έχουν αναφερθεί τα οποία δεν ωφελούν, είναι πάρα πολύ βασικό να συμμορφωθεί το Μπουρούντι και να απελευθερωθεί ο κύριος Ρογκούρικα αλλιώς θα πρέπει δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας Κοτονού να ανασταλεί η χορήγηση αυτής της ενίσχυσης προς το Μπουρούντι. Ευχαριστώ. Ο επόμενος συντάκτης Ιγνασίου Κογκρά επίσης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Ρογκούρικα ε, έχει αυτό το, το ραδιοφωνικό σταθμό και πέραν των όσων λέει ε, ε, το, το κράτος είχαμε ε, την αποτρόπη μεταχείριση φόνο διβιασμού αυτών των τριών καλογριών και το οποίο τα απεκάλυψε οπότε κατεπατήθη η ελευθερία του τύπου όμως θα πρέπει να δούμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει όλη την οικονομική βοήθεια στις εκλογές που θα ακολουθήσουν στην χώρα και επομένως φυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος επειδή δυσκόλεψε σε δύσκολη θέση τέλο πάντων την κυβέρνηση. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη χώρα αυτή. Να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση του Ρόμπουλ Γκουρικα με το ψήφισμα. Ευχαριστώ και η κυρία Σέντρα Ροντρίγκε, επίσης ε, συντάκτης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή μας στο θέμα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι. Ζητάμε την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και του εκφράζεστε και πετούμε και ελευθερία για τον Μπόμπο Ρουγκουρίγκα. Θέλουμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή του κόσμου και στο γεγονός ότι το Μπουρούντι είναι από τις 10 πιο φτωχές χώρες του κόσμου και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι οι δυτικές δυνάμεις έχουν ε, μεγάλες ευθύνες για την ακραυτή ε, φτώχεια στην περιοχή αυτή της Αφρικής. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι έχει καφέ, έχει μπαμπάκι, έχει κοβάλτιο, έχει χαλκό, νερό, ένα σωρό ε, πόρους. Περιμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις χώρες μέλη να στηρίξουν τη χώρα για να αντιμετωπίσει την χρόνια, το χρόνιο λοιμό και για να ενισχυθεί η τοπική γεωργία και η οικογενειακή γεωργία που είναι ε, βασικό έσοδο για την χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιώζεφ Βάιντχολτσερ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι τα, τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν φοβερές εξελίξεις στο Μπουρούντι. Σε αυτή τη δοκιμαζόμενη χώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πως το καλύτερο μέλλον περνάει μόνο μέσα από ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εκλογές που έρχονται θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως για αυτό να υπάρχει ελευθερία τύπου. Όσο πιο κοντά έρχονται οι εκλογές, τόσο πιο πολύ μειώνονται τα περιθώρια. Ο Μπόμπο Ρουγκουρίκα είναι μια σημαντική φωνή για την δημοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν να αφαιθεί αμέσω και ανεφόρον ελεύθερος. Πρέπει και εμείς να προσθέσουμε τη φωνή μας στην πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Μωρίς Πόγκα, τελευταίος των συντακτών, για ένα λεπτό επίσης. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η δεύτερη φορά από την αρχή αυτή τη θητεία που το Κοινοβούλιο μα ζητάει από την κυβέρνηση του Μπουρούντι να τηρήσει τι υποχρεώσει του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα έχουμε τον κύριο Μπομπ Ρουγκουρίκα που μα απασχολεί. Κρατείται από τι 20 Ιανουαρίου στη φυλακή επειδή έθεσε υποφεσβήτηση την κυβέρνηση όσον αφορά τη δολοφονία των τριών Ιταλίδων μοναχών, λέγοντας ότι υπήρχε συμμετοχή στη δολοφονία των μυστικών υπηρεσιών. Και επειδή δεν θέλησε να πει ποια ήταν η πηγή του, ο κύριος Ρουκούρικα βρέθηκε 20 χρόνια στη φυλακή με διάφορες κατηγορίες μεταξύ άλλων έλλειψη ελληνικής κτλ. Εμείς ζητάμε την απελευθέρωσή του άνευ όρων. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα πλησιάζουν οι εκλογές τον Μάιο που μας έρχεται. Είναι θέμα αξιοπιστίας το, της ίδιας της των εκλογών αυτών. Αυτό διακυδεύεται. Ευχαριστούμε κύριε τους Πόσπισιλ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντάκτες της πρότασης αυτής ψηφίσματος. Εγώ πιστεύω ότι η υπόθεση του κύριου Ρουγκούρικα είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι άλλη μια περίπτωση δημοσιογράφου ο οποίος κατηγορήθηκε επειδή ερευνούσε, επειδή έκανε τη δουλειά του. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η κατάσταση μάλιστα είναι ακόμα χειρότερη επειδή κατηγορήθηκε ο ίδιος τελικά ότι συνεργάστηκε με το, για το έγκλημα αυτό. Πρόκειται δηλαδή για μια φοβερή κατάχρηση που γίνεται παραβίαση της δικαιοσύνης της ίδιας. Σαφέστατα λοιπόν το καταδικάζουμε. Το Μπορούντι είναι τέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη χώρα αυτή οικονομικά. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να ζητάμε μόνο την άμεση απελευθέρωσή του, αλλά και την διερεύνηση του εγκλήματος κατά τριών Ιταλίδων μοναχών που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν γίνει η έρευνα αυτή θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις κατά τις χώρες. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά κύριε Σκαπούτο. Μόλις πριν εβδομα... λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές είδαμε τι έγινε ε, στο Μπουρούντι που είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ε, διαφθορά είναι πεντηκοσιωστή εβδομή θέση σύμφωνα με τις διεθνείς φορείς οπότε βλέπουμε το, τι, έγινε ε, με αυτή την περίπτωση του Μπόμπρου Γκουρίκα που έχει ε, αυτό το σταθμό τον ραδιοφωνικό έκανε δημοσιογραφική έρευνα όσον αφορά τις τρεις ιεραποστόλες της Ιταλίδες οπότε βλέπουμε ότι ε, υπέστησαν βασανιστήρια σωματικά και ψυχολογικά έχουν κινητοποιηθεί ε, οι Εθνείς Χωρίς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αρνήθηκαν οι αρχές να τον αποφυλακίσουν. Θα πρέπει αποφασιστικά κάτι να κάνει η Ευρώπη, να κάνει ένα διάβημα και να απαιτήσει από τις αρχές την απελευθέρωσή του. Και έτσι να ισχύει δημοκρατία στην χώρα. Καστάλντο ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσο κοστίζει σε κάποιον η έρευνα της αλήθειας πόσο θα πρέπει να πληρώσει. Είχαμε αυτές τις τρεις καλόγριες. Η Μπερναρδέτα, η Όλγα και η Λουκία το πλήρωσαν με την ζωή τους. Και ο ακτιβιστής αυτός, ο κ. Ζουγκουρίκα, τώρα θα πληρώσει το ότι ήθελε να διασκεδάσει τις αμφιβολίες, να, να βρει την αλήθεια με 20 έτη κάθερξης. Τον πήγανε σε κάποια πολύ σκληρή φυλακή τώρα εκεί βοηθά και είναι πολύ άνετο αυτό η κυβέρνηση το να φυλακίζει κάποιους που την κάνουν να αισθάνεται δύσκολα. Οπότε θα πρέπει να απαιτηθεί η αποφυλάκηση και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Κάτι το οποίο αφορά κάθε δημοσιογράφο και κάθε ακτιβιστή που παλεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, έχουμε επομένω τώρα αυτές τις εκλογές σε αυτή τη χώρα που φημώνει δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει κάτι τέτοιο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γκάμπουσα ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο πράγματι, γιατί για τον Μπουρούντι έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ μέχρι τώρα. Στι 20 Ιανουαρίου φυλακίστηκε λοιπόν ο κύριο Ρουκούρικα από το Αφρικανικό Ραδιόφωνο, επειδή είχε κάποια ρεπορτάζ για τη δολοφονία αυτή των τριών Ιταλίδων μοναχών που πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και στήριζαν την τοπική κοινότητα. Αναφίβολα είναι κάτι πολύ ανησυχητικό αυτό. Ανησυχητικό ω αυτό αλλά και εξαιτία τη ε, τιμωρία ε, που επευλήθη στον κύριο Ρουγκουρίκα, ο οποίος με λάθο κατηγορία μπορεί να φτάσει 20 χρόνια στη φυλακή. Οφείλουμε λοιπόν να ζητήσουμε από τις αρχές του Μπουρούντι την άμεση απελευθέρωση του κύριου Ρουγκουρίκα, γιατί η κράτησή του αποτελεί περιορισμό δυσανάλογο περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης και να ζητήσουμε από τον Τουρούντι να τηρήσει τις συμφωνίες που έχει υπογράψει μαζί μας ή ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα ή αυταρχισμός και καταδίκη. Ευχαριστούμε. Τα Μπαρντέλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία έκφρασης είναι θεμέλιος λήθος της δημοκρατίας. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στο Μπουρούντι καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του Μαΐου είναι πραγματικά τρομερό. Μιλάμε για την περιοχή των μεγάλων λιμνών της Αφρικής, ε, μια σημαντική περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσει τον λαό του Μπουρούντι, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του και να υπάρχει ελευθεροτυπία και ένα σταθερό περιβάλλον και να συνεχίσει την πορεία του προς την δημοκρατία. Η Ευρώπη πρέπει να φροντίσει να μην υπάρξει οπισθοχώρηση. Οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση του Μπορούντι να σεβαστεί τι δεσμεύσει, τη, να οργανώσει σωστέ εκλογέ να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ε, όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στι υφιστάμενε συμφωνίε. Ζητώ την άμεση απελευθέρωση του κυρίου Ρουγκουρικά. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε τέσσερις που ζήτησαν το λόγο. Θα μιλήσουν όλοι κύριος ε, Βάντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Μπομπρουγκρικα ήταν διοκτήτης ενός σταθμού και συνελήφθη όταν δημοσίευσε ρεπορτάζ σε σχέση με την ανθρωποκτονία των τριών Ιταλών, Ιταλίδων Ιεραποστόλων. Πρόκειται για μια χώρα όπου διώκονται οι ακτιβιστές. Απαγορεύεται η επίκριση της κυβέρνησης. Είπαμε και γιατί έγινε και με τον Δ. Μπονίμπη. Όμως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να σεβαστεί την ελευθερία του τύπου και να συμμορφωθεί με την Συμφωνία Κοτονού γενικότερα. Οι... Τώρα θέλουν να καταδικάσουν τον κύριο Γκρίγκα και αυτό θα πρέπει και εμείς να το επικρίνουμε γιατί θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή και αυτό να θεωρηθεί προϋπόθεση ούτως ώστε να θεωρηθούν νόμιες εκλογές της χώρας. κυρία Κέγγε για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακόμα μια σύλληψη, ακόμα μια καταπάτηση της ελευθερίας έκφρασης που πλήσει και τους δημοσιογράφους και τους ακτιβιστές και την ε, αντιπολίτευση στη χώρα. Για άλλη μια φορά έχουμε μια τέτοια περίπτωση όπως την περίπτωση Μπονίμπο που είχαμε ε, καταδικαστά πράγματα επιδεινώνεται και θα έχουν και τις προεδρικές εκλογές. Τον ε, κατηγόρησαν ότι ήθελε να, να ρίξει φως όσον αφορά την ανθρωποκτονία ε, των τριών αυτών ε, ιεραποστόλων, οπότε θα πρέπει να γίνουν σε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης. Να ισχύσει η ρήτρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων της Συμφωνίας Κοτονού για τα δημοκρατικά δικαιώματα και αυτό προβλέπεται επίσης και στον ε, στον, στην χάρτα δικαιωμάτων που ισχύει για την Αφρική οπότε θα πρέπει αυτή η ρήτρα να εφαρμοστεί και να καταδικάσουμε κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση σε όλη την προκλήκη περίοδο ούτω ώστε να μην επαναληφθούν οι ε, καταπατήσεις των δικαιωμάτων να υπάρξει εκδημοκρατισμός, ασφάλεια και ειρήνη στον Μπουρούντι και σε όλη την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Κύριος Μαριάς, ένα λεπτό. Πρόεδρε, η παρα δικαιωμάτων εντείνεται το τελευταίο διάστημα στο μπουρούντι. καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές και γενικές εκλογές εντός του 2015 το καθεστώς εντείνει τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο της ελευθερίας του τύπου. ταυτόχρονα περιορίζει τους όρους άσκησης της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. πρόσφατα κατάδειλη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μπουρούντι αποτελεί παράνομη σύλληψη και προφυλάκηση του γνωστού ακτιβιστή και διευθυντή ραδιοφωνικού σταθμού μπομπ ρουγκουρίκα διότι τόλμησε με τεκμηριωμένο ρεπορτάζ να ασχοληθεί και να αποκαλύψει τα της δολοφονίας το σεπτέμβριο του 2014 τριών Ιταλίδων καλογρεών. Στηρίζουμε λοιπόν το ψήφισμα που καταδικάζει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι και ζητούμε την άμεση αποφυλάκηση του ακτιβιστή Μπομπ Ρουγκουρίκα. Ευχαριστώ. Ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι κοινό έχουν ο Ρουγκουρίκα και ο Μπανταούι. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι παράνομα κρατούνται, έχουν φυλακιστεί αδίκως, χωρίς λόγο. Έχουμε να κάνουμε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω εδώ για θέματα αυτά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, γιατί πρέπει να ακουστεί αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε πρόβλημα να καταδικάζουμε τέτοιες παραβιάσεις όπου και να συμβαίνουν και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε σαν να έχουν να κάνουμε ένα και μόνο άτομο. Το Φεβρουάριο έχουμε ένα χρόνο από τις διαδηλώσεις της Βενεζουέλα που με βία σταμάτησαν και οδήγησαν σε φυλάκιση εκατοντάδων ανθρώπων. Ο Λόπεθ, για παράδειγμα, εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή και εμεί έχουμε ζητήσει επανελειμμένω να ελευθερωθεί. Και αυτό λοιπόν μαζί με του άλλου αδίκω έχει καταδικαστεί. Εδώ πρέπει να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε. Τουρκάι. Ένα λεπτό. Τουρκάης. Mm. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς το Μπουρούντι, όπως το ακούσαμε, δεν ε, τηρούνται. Δεν γίνεται, υπάρχει σεβασμός ούτε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε της ελεύθερης έκφρασης, ούτε της ελευθερίας του τύπου. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουμε καταδικάσει εδώ στο σώμα όπως το υπενθύμησε και συνάδελφος και αυτά που συμβαίνουν για παράδειγμα στη Βενεζουέλα. Οι διώξεις και οι φυλακίσεις δημοσιογράφων όπου και αν λαμβάνουν χώρα είναι μια κατάφορη παραβίαση, όπως το υπενθύμησαν και συνάδελφοι, ιδίως τώρα που το Μπουρούντι βρίσκεται λίγο πριν τις εκλογές. Οι εκτιβιστές, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στη φυλακή παράνομα στο Μπουρούντι πρέπει να ελευθερωθούν. Πρέπει να ισχύσουν δημοκρατικοί κανόνες και σε αυτή την Αφρικανική χώρα. Και αποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να επενθυμίσω σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται υποκράτηση αλλού στον πλανήτη Γη, ότι και γι' αυτούς ζητάμε να ελευθερωθούν αμέσως όπως και ο Λόπεθ στην Βενεζουέλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γιάφκοφτσιτς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σήμερα συζητούμε για άλλη μια φορά με τον κλασικό τρόπο. Έχουμε εδώ ένα αποτρόπιο έγκλημα. Έχουμε συμφέροντα στην περιοχή των μεγάλων λιμνών και έχουμε επίσης και τη Συμφωνία Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόκειται για ακόμα μια φορά για έναν δημοσιογράφο. Ανέκαθεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούσαμε για τέτοιες περιπτώσεις. Για τέτοια εγκλήματα. Επίσης τα, λέμε και για το Κονγκό και πολύ συχνά για τις ε, μεγάλες λίμνες αυτή την περιοχή. Μιλούμε για θεμελιώδεις ελευθερίες, αλλά χρειάζεται μια κοινή πολιτική. Θα πρέπει να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι με όλους τους εταίρους μας, να τους εξηγήσουμε ότι θα πρέπει να σεβαστούν στο ελάχιστο κάποια βασικά άνθρωπινα δικαιώματα. Να μια οριστική θέση. Φαρία, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η υπεράσπιση της ελευθερίας ε, της έκφρασης ε, και του διαχωρισμού κράτους εκκλησίας οδήγησε στην δεκαετή φυλάκιση του Ραϊφ Μπαντάουι και την τακτική μαστίγωσή του. Ο βασιλιάς Αμπτουλάχ ε, Αναμένεται να του δώσει χάρη, αλλά προς στιγμή δεν ε, γίνεται τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παραπέμψω στο ερώτημα της 4 Φεβρουαρίου που υπέβαλα μαζί με άλλους ε, ευρωβουλευτές στην κυρία Μογκερίνη. Το ερώτημα ήταν τι, με, τι θα κάνετε για να ασκήσετε πίεση στην ε, Σαουδική Αραβία να αναθεωρήσει τον ποινικό της κώδικα. Ε, ευχαριστώ. Έχω λάβει Με συγχωρείτε λάθος μου, λέει ο πρόεδρος. Όλοι, όλοι θέλουμε να τελειώσουμε νωρίτερα, λέει ο επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Είμαι ευγνώμων στους βουλευτές που τόνισαν το θέμα αυτό. Υπενθυμίζω πως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Μπουρούντι το Σεπτέμβριο βοήθησε στην απελευθέρωση με εγγύηση του κυρίου Πιέρ Κλαβέ Μπονίμπα. Επίσης ενθάρρυνε έναν πιο εντατικό πολιτικό διάλογο με την Μπουζουμπούρα. Παρόλα αυτά έχουμε σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επιγόντως καθώς πλησιάζουν ε, βουλευτικές και προεδρικές και δημοτικές εκλογές. Να τονίσω την ανησυχία την δικιά μου και της κυρίας Μογκερίνη για την σύλληψη του Μπομπ Ρουγκουρίκα. Αυτό έλαβε χώρα μετά την εκπομπή του που ανέφερε ε, την δολοφονία τριών ε, Ιταλίδων καλογρεών ε, η οποία δολοφονία βεβαίως πρέπει να διαρευνηθεί. Γύρονται λοιπόν σοβαρές ε, ανησυχίες δεδομένου και του πολιτικού κλίματος. Οι κατηγορίες εναντίον του μοιάζουν δυσανάλογες και δεν υπάρχει νομική βάση για την κράτησή του. Το ζήτημα θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του νόμου περί μίμιε της χώρας ή μέσω του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στην Μπουζουμπούρα επισκέπτονται τακτικά τον κύριο Ρουγκουρίκα στη φυλακή για να δουν τις συνθήκες κράτησής του. Θα παρακολουθήσουμε την υπόθεσή του και θα ζητήσουμε σεβασμό της ε, ελευθεροτυπίας. Λίγο μετά την σύλληψη του κυρίου Ρουγκουρίκα η υπόθεσή του ετέθη ως ζήτημα στον διάλογο που έχουν οι επικεφαλείς της αντιπροσωπείας της Ένωσης με τις αρχές του Μπουρούντι επέμειναν στον σεβασμό της νομιμότητας και του νόμου περί ελευθεροτυπίας και ελεύθερης έκφρασης ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή του. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Τα μηνύματα αυτά δημοσιοποιήθηκαν και σε ένα ανακοινοθέν. Επίσης εξέφρασαν ανησυχία για τον πιθανό πολιτικό αντίκτυπο της υπόθεσης αυτής καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά το πολιτικό κλίμα και η αξιοπιστία των αρχών και η εκλογική διαδικασία. Έχοντας αυτά κατά νου, επαναβεβαιώνω την σημασία που έχει για μας οι εκλογές αυτές να είναι διαφανείς, ειρηνικές και αξιόπιστες με τη συμμετοχή όλων Η κράτηση του Μπομπ Ρουγκουρίκα στέλνει ένα ανησυχητικό μήνυμα για τους δημοσιογράφους στον Μπουρούντι. Καλωσορίζω το ότι επικοινωνούμε τακτικά με τους ε, ομολόγους μας ε, του Μπουρούντι στον πολιτικό διάλογο και έτσι έχουμε μια επαφή σε επίπεδο θεσμικό στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχουμε υπογράψει και βεβαίω υπογραμμίζουμε πως η στήριξή μας στις εκλογές εξαρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μπουρούντι μεταξύ των οποίων και αυτές που έχουν αναλυφθεί για τον εκλογικό νόμο και τον οδικό χάρτη και οπωσδήποτε θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία να Ε, παρακολουθήσουμε την υπόθεση Ρουγκουρίκα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε.